είναι εδώ η συζήτηση, προφορεί αύριο στι 12. Σας ευχαριστώ. Και περνούμε τώρα στο προσεχές θέμα της ημερησία διάταξης. Που είναι η έκθεση του κύριου Κάρενς. Διακυβερνητικέ συμφωνίε που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα τη ενέργεια. Διερωτώ με όμω αν εκ Επιτροπή παραμένει ο κ. Δεχούχτ στην αίθουσα. Όχι. Ο κύριος Έτσιγκερ. Καλώς ήρθατε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πιστεύω σε ένα-δύο λεπτά, δευτερόλεπτα, μόλις καθίσει ο κύριος Επίτροπος. Ξεκινούμε λοιπόν με τέσσερα λεπτά για τον εισηγητή. Κύριο Κάρενς, έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Στο δέτο τομέα του φυσικού αερίου έχουμε Ξανόμενε τάσει σε μια εξάρτηση τη τάξη του 60%. Στον τομέα του πετρελαίου έχουμε εξάρτηση κατά 80% και περισσότερο. Για μας βεβαίω στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, ασφαλείς ε, προμήθειες ενέργειας. Αλλά η κατάσταση ποια είναι σήμερα. Η κατάσταση σήμερα είναι ότι κάθε κράτο μέλο ε, συνάπτει διμερεί συμφωνίε με τρίτε χώρε, χώρε προμηθευτέ δηλαδή, για την ε, προμήθεια ενέργεια. Συμφωνίε οι οποίε ε, δεν είναι διαφανεί, δεν γνωρίζει κανεί τι περιλαμβάνουν. Πέραν του κράτους μέλους που τις έχει συνάψει βεβαίως. Και έτσι μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία στο θέμα αυτό. Υπάρχει ανταγωνισμός ως προς τη χρήση των οδών ε, προμήθειας και όπως είπα διαφανείς εμπορικές σχέσεις και το πρόβλημα είναι ότι για μας τον καταναλωτή είναι πολύ πιο ε, υψηλέ οι τιμές ε, γιατί δεν λειτουργεί όπως πρέπει ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει ευρωπαϊκό συντονισμός δεν υπάρχει διαφάνεια και έτσι θα έλεγα με την αρχή του διέρη και βασίλευε, η κάθε χώρα χωριστά δηλαδή συνάπτει σχέσεις, ε, ταλαιπωρείται περισσότερο ο καταναλωτής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του του 2011 ανέφερε την πρόταση να ε, δώσει επιτροπή λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Αυτό λοιπόν προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις προτάσεις αυτές συζητούμε σήμερα και για να σας ε, δώσω με απλά λόγια να καταλάβετε, η πρόταση είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όπου τα κράτη-μέλη θα ε, χορηγούν τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις σχετικές με τις διμερείς σχέσεις που έχουν, τις διμερείς συμφωνίες, τις οποίες ε, πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να τις αξιολογεί και να ελέγχει κατά πόσον ε, συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κυρίως νομοθεσία σχετικά, σχετική με τον ανταγωνισμό και στη συνέχεια με ένα συντονιστικό μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αρχίσει να ομιλεί με μία, μία ενιαία φωνή ε, στις επαφές της με τους προμηθευτές ενέργειας. Εμείς στην Επιτροπή μας Συστώντα το θέμα αυτό, συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί και 90% των μελών της Επιτροπής ε, βιομηχανία, έρευνα και ενέργεια υποστήριξαν την ε, πρόταση αυτή. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εντολή λοιπόν για ένα τριμερή διάλογο. Μέχρι που ήρθε η ώρα να γίνει αυτός ο διάλογος με, τον, ε, με τους κοιόδης όπου ε, επήλθε η ρήξη για το Συμβούλιο δεν θέλει να συζητήσει τέτοιες προτάσεις. Η Δανική Προεδρία σε τρεις τέτοιους τριμερείς διαλόγους βοήθησε στην επιτεύξη μιας συμβαστικής λύσης αποδεκτής για το Κοινοβούλιο αλλά και για το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία, η οποία λύση έχει ως εξής. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών στον οποίο θα τροφοδοτούμε όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τις ε, αλλά και τι συμφωνίες τους στα κράτη-μέλη και έτσι η Επιτροπή θα μπορεί να δει μέσα από αυτό το παρατηρητήριο τα στοιχεία τα σχετικά με αυτές τις συμφωνίες και ταυτόχρονα οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνει θα, την επιτρέ... θα τις επιτρέπουν να έχει μια πιο ισχυρή θέση στη διαπραγματεύσεις με τα τρίτα κράτη. Δεν θα μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει σε μια προκαταρκτική φάση αυτής της διαδικασίας. Γιατί αυτό δεν το δέχτηκε το Συμβούλιο. Πλην όμως, εγώ θα ζητούσα από τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την πρόταση αυτή, έστω και αν δεν είναι 100% αποδεκτή, διότι πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι κατά μια ε, πρόσμια, μάλλον αποδεκτή ενεργειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βήμα το βήμα μια ενεργειακή πολιτική, η οποία θα είναι θετική για του καταναλωτέ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, και παρακαλώ τον Επίτροπο κύριο Έτσιγκερ να λάβει το λόγο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το ζήτημα μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής κοινοτικής θέσης στο θέμα της ενέργειας. Συμφωνώ βεβαίως με τον ε, κύριο Καρίνς. Περιέγραψε την όλη διαδικασία και την πορεία μέχρι τώρα και μας είπε ότι μπορέσαμε να έχουμε μια καλή, καλά συντονισμένη και επιτυχή εν τέλει διπλωματική προσπάθεια συντονισμού στην υπόθεση αυτή. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Μπορεί να έχουμε συμφωνίες κρατικές με κράτη τρίτα, τα οποία, οι οποίες συμφωνίες ίσως να μην ε, εγγράφονται, να μην είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο που όμως συνάπτονται από τις χώρες μέλη, γίνονται δεκτές δηλαδή από τις τρίτες μέλη, όχι γιατί θέλουν να, κάνουν, ε, να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί βρίσκονται υποπίες σε σχέση με τα τρίτα κράτη προμηθευτές. Άρα λοιπόν, η δημοσιοποίηση αυτών των συνθήκων, αυτών των συμφωνιών είναι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίζουμε, να ελέγξουμε, να επαληθεύουμε αν όντω είναι συμβατές αυτέ οι συμφωνίε με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αν δεν είναι να κοιτάξουμε να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να τι τροποποιήσουμε. Επίση, δεύτερον, με την πρόταση αυτή προκύπτουν ε, πλεονεκτήματα για τον ανταγωνισμό όπω και μειονεκτήματα όμω. Γιατί εάν γνωρίζει το τρίτο κράτο, όλε τις συμφωνίε που έχει συνάψει αλλά τα ευρωπαϊκά κράτη μόνο το καθένα τη δική του ε, συμφωνία προφανώς ε, μόνο με διαφάνεια περισσότερη μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση μα. Επίσης αυτό μπορεί να ενδιαφέρει και τον επενδυτή στον ιδιώτη επενδυτή σε ένα δίκτυο υποδομών για τη μεταφορά των ενεργειακών αυτών πηγών. Οι διακρατικές ε, αυτές σχέσεις επίσης μπορεί να προξενήσουν προβλήματα στην ασφάλεια δικαίου αν δεν είναι γνωστές διαφάνεια και η επαλήθευση της συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο μας προστατεύουν από δυσάρεστες εκπλήξεις, από προσφυγές για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από διαδικασίες οι οποίες μπορεί να θέσουν ένα αμφιβόλο και κάποιες επενδυτικές προσπάθειες. Και έτσι προχωρώ στα, ε, στις ελλείψεις σχέση με αυτά που είχαμε και εμείς επιδιώξει αλλά και το Κοινοβούλιο ζητήσει ως προς τη συμφωνία αυτή, ως προς τη ε, συμβαστική αυτή λύση γιατί υπολείπεται σε σχέση με αυτά που είχαμε προτείνει. Σημειώνω όμως ότι πρόκειται για μια ιστορική πρωτιά γιατί είναι η πρώτη φορά που συζητούμε μια, ένα πρώτο βήμα μια κοινή ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τρίτα κράτη που πια δεν μπορούν τόσο εύκολα και τόσο απλά να επιβάλλουν τους όρους τους. Στην ε, πρόταση έχουμε όλα τα στοιχεία, δηλαδή έχουμε την υποχρέωση να κατατεθούν, να δημοσιοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες ενεργειακές συμφωνίες στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει και ως παρατηρητής στις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας αυτές και να δώσει συμβουλές της. Υπάρχει δυνατότητα και η παράκληση να είναι συμβατές αυτές οι συμφωνίες με ε, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και να επαληθευτεί η συμβατότητα των ήδη συναυθισών συμφωνιών με το κοινοτικό δίκαιο. Όλα αυτά ενισχύουν λοιπόν την εσωτερική αγορά, όλα αυτά ενισχύουν τη θέση των κρατών μελών σε σχέση με τα τρίτα κράτη προμηθευτές. Και έτσι, θεσπίζοντας αυτή την ε, συμφωνία, νομοθετώντας την δηλαδή, μπορούμε να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερως. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει η επακριβής επιτήρηση και η τήρηση των νέων αυτών νομοθετημάτων και των διατάξεων μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να επαληθευτεί με προσοχή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει την επιτήρηση του κατά πόσον υπάρχουν επαρκή μέσα, όργανα στη διάθεσή μας και αν όχι θα φροντίσουμε την επόμενη χρονιά να καταθέσουμε μια νέα πρόταση για την ενεργειακή πολιτική που πιστεύω θα αποτελέσει ένα σημαντικό και νέο βήμα αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να δούμε εάν χρειάζεται ένα επιπλέον βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κυρία Γιαννάκου, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα αυξήσει de facto τη συνέπεια και τη συνοχή των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων της Ένωσης, ενισχύοντας παράλληλα και τη στρατηγική θέση της Ένωσης στη σχέση με τρίτες χώρες. Σήμερα παρεμβαίνω ως εκπρόσωπος και εισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ευρωπαϊκή ένωση συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ενέργειας καθιστώντας επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις τη λειτουργία και τον ενεργειακό εφοδιασμό της αγοράς ενέργειας. ο νέος μηχανισμός αυτός πράγματι μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη διαπραγματευτική δύναμη των κρατών μελών μέσω της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της εμπειρογνωμοσύνης της επιτροπής όσο αφορά στο κοινοτικό δίκαιο ταυτόχρονα η ασφάλεια δικαίου που θα προκύψει για τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις μέσω ενός σταθερού νομικού πλαισίου θα καταστήσει ευκολότερη τη χρηματοδότηση σχετικών έργων από την ένωση και μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιταχύνει το χρόνο υλοποίησης. σαφέστατα ο καλύτερο συντονισμό που μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτού του μηχανισμού δεν πρέπει να ερμηνευθεί ω μικρότερη ευελιξία στα κράτη μέλη. το όλο εγχείρημα θα έχει επικουρικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα κράτη μέλη ω αρμοδίους Σύναψη ενεργειακών συμφωνιών με τρίτες χώρες. η εμπλοκή όμως της επιτροπής μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά ωφέλη συνδράμοντας ουσιαστικά τα κράτη μέλη ιδιαίτερα κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους συμφωνιών. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Thank you very much, Madam Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιαννάκου. Τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Ζαντό από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Οπότε θα περάσουμε στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Καστίγιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καρίν στον εισηγητή και όλους τους κοιόδης που μαζί του που από κοινού αποφάσισαν να προχωρήσουν με αυτές τις διαπραγματεύσεις μέσα στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων όπου συναντήθηκαν δυσκολίες, όπως μας είπε και ο κύριος Καρίνς. Επειδή έγινε αυτή η κοινή ε, προσπάθεια με αποφασιστικότητα, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά θα υπάρξει μία ανταλλαγή πληροφοριών και ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ κρατών μελών και ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις διακυβερνητικές συμφωνίες ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό. Έτσι θα υπάρχει ε, μία χαρτογράφηση των δικτύων εφοδιασμού και θα μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τη προμήθεια, την προμήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία τι κάνουμε. Βρισκόμαστε στην οδόστρωση ανοίγοντας ένα νέο δρόμο για να μπορέσουμε να δώσουμε άλλη ταχύτητα και να προχωρήσουμε με σπουδή στη, στον ενεργειακό εφοδιασμό. Εάν δεν γίνει, αν δεν ανοίξει αυτός ο δρόμος, τότε χάνουμε μία χρυσή ευκαιρία. Θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά με, μεγάλο χρονικό, με μεγάλη χρονική απόσταση. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ του, τον εισηγητή και τους σκιώδης. Σας ευχαριστούμε γιατί κρατήσατε και το χρόνο σας. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών και δημοκρατών ο κύριος Λάγκια για τρία λεπτά. Κύριε Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Σίγητα, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Σιγητή για τη δουλειά του και πάνω απ' όλα για την υπομονή που έδειξε σε αυτές τις ε, μήνυ διαπραγματεύσεις. Και κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόταση αλλά και γενικότερα για τη δουλειά που κάνετε στον τομέα της ενέργειας που είναι πολύ καλή. Δυστυχώς αυτός που θα έχω να επικρίνω σήμερα δεν είναι παρόν, το Συμβούλιο δηλαδή. Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα το πω ξεκάθαρα, έχω ζήσει περίπου 50 διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου, συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο αλλά πρώτη φορά είδα το Συμβούλιο να εκβιάζει ουσιαστικά με τη συμπεριφορά του το Κοινοβούλιο και να λέει ή αυτό ή τίποτα. Ούτε είχα δει ποτέ το Συμβούλιο να συμπεριφέρεται με τόσο αρνητικό τρόπο σε διαπραγματεύσει τριμερούς διαλόγου. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, όταν ακούμε τα ωραία κηρύγματα για πιο πολύ Ευρώπη, όπως και σήμερα το πρωί, και που συζητούμε όλη αυτή την περισσότερη Ευρώπη που χρειαζόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και συνεννόηση για την πολιτική μας, για την ενέργεια και εσείς το είπατε κύριε Επίτροπε, η ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη και για την οικονομική της ανάπτυξη και για το μέλλον και για τον προσδιορισμό της, των προοπτικών της μηχανικής μας πολιτικής της σημασίας. Και γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή πολιτική κυρίες και κύριοι μπορεί να διαμορφωθεί μόνο εφόσον έχουμε συνεννοηθεί εμείς μεταξύ μας για μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική μέσω των συμφωνιών μας με τα τρίτα κράτη. Στο βαθμό αυτό λοιπόν και με όλη την κατανόηση που μπορούμε να δείξουμε. και την κατανόηση ότι δεν θέλουν όλοι να έχουν παρά μόνο ένα κοινό, ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Πρέπει, πρέπει να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα υποχρεωτικά για να μπορεί η Επιτροπή να συμμετέχει έστω και ω παρατηρήτρια σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Αυτό το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε για να έχουμε μια εξωτερική πολιτική για την ενέργεια στην πράξη, μια ουσιαστική πολιτική η οποία δεν υπάρχει μέχρι τώρα γιατί δεν την επιτρέπουν τα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν αύριο με τις τροπολογίες και την υποστήριξή σας να μπορέσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο να δεχθεί τις θέσεις μας. Και κύριε Επίτροπε, Ελπίζω αυτό το οποίο αναφέρατε και προς το τέλος ε, της ομιλίας σας να το υλοποιήσετε πράγματι, δηλαδή την επαλήθευση τη συμπεριφορά του Συμβουλίου στο μέλλον, έτσι ώστε πράγματι ε, όταν έρθει η ώρα να γίνει και μια πραγματική μεταρρύθμιση της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λάγκα και τώρα ακολουθεί ο κύριος Κρόιτσμαν για 1,5 λεπτό. Κύριε Επίτροπε αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πολλούς τομείς ε, πολιτικής γίνεται λόγος ε, σε εθνικό επίπεδο, για εθνικό επίπεδο ή για ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεννόηση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αυτή η για ευρωπαικο επιπεδο και στην ενώση δυστυχως ομως ευρωπαϊκή στην ενεργειακή πολιτική μας με τις τρίτες χώρες και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη φιλόδοξη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, τα, και αντιμετωπίζουν ε, την άρνηση, την αρνητική στάση των μελών του Συμβουλίου των κρατών μελών δηλαδή. Δεν υπάρχει μια κοινή ενεργειακή εξωτερική πολιτική, αλλά θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε τις ε, απαντήσεις, να δώσουμε τις απαντήσεις για να έχουμε μια ε, ενεργεία που μπορούμε να πληρώσουμε να είναι υπερβολικά ακριβή όταν ε, η παγκοσμιοποίηση και οι κύριοι παράγοντες στην αγορά της ενέργειας μας επιβάλλουν τους όρους, πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε. Η κοινοβουλευτική μας λοιπόν ε, θέση ήταν εξ αρχής γνωστή. Πρέπει να υπολογίσουμε ότι θα υπάρξουν αντιστάσεις το Συμβούλιο δεν έχει περιθώριο για διαπραγματεύσει, δεν αφήνει μάλλον περιθώριο για διαπραγματεύσει, μα ε, βάζει όλου σε σκέψει και θα πρέπει να αξιολογήσουμε τι επιλογέ γιατί μπορούμε επιτέλους, έχουμε μια ευκαιρία να προσδιορίσουμε ένα πλαίσιο συνεννόησης το οποίο μπορεί να μας καθοδηγήσει στα επόμενα χρόνια καλύτερο, έστω και με τις ελλείψεις του, από το να μην ε, είχαμε καμία συμφωνία και θα, να έπρεπε δηλαδή να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Έτσι λοιπόν εγώ θα πρότεινα να καταψηφιστούν οι τροπολογίες των σοσιαλιστών και δημοκρατών και θα ήθελα θερμά και ρητά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αγωνιστική του διάθεση και για τις προσπάθειές του να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε για ένα λεπτό. E, e, Κυρίες και κύριοι, μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά του φυσικού αερίου δεν είναι και πολύ δημοφιλή σε ορισμένες χώρες. Τα τελευταία χρόνια η δίκαιη πρόσβαση στα δίκτυα διανομής και στις εξαγωγές φυσικού αερίου είναι κάτι το οποίο έχει αμφισβητηθεί ανοιχτά από τη Ρωσία η οποία εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Gazprom θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Παρ' όλα αυτά όμως σαν μονοπωλιακή κρατική εταιρεία προστατεύει την θέση της. Και λόγω του ότι η αγορά στην κεντρική Ευρώπη δεν είναι σωστά αναπτυγμένη, επιβάλλει η Gazprom τελικά άδικες τιμές, υπερβολικές τιμές και απαράδεκτους κανόνες. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες βελτίωσης του ανταγωνισμού δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις αρχές όμως της κοινή αγοράς. Πριν μερικούς μήνες ενισχύσαμε την προστασία της αγοράς φυσικού αερίου με τον έλεγχο μηχανισμό των συμφωνιών αυτών των επιμέρους. Νομίζω ότι δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που κάναμε και με τον εισηγητή την ευκαιρία αυτή τελικά τη χάσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σιμάνσκι. Κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ε, κύριοι συνάδελφοι η έκθεση κάριν έρχεται πράγματι να επιλύσει πολλά προβλήματα στην ενεργειακή πραγματικότητα της ευρώπης. για παράδειγμα αυτή την περίοδο έχουμε την περίπτωση του ενεργειακού εφοδιασμού της λιθουανίας για την οποία περίπτωση η επιτροπή έχει διατάξει έρευνα έχει διεξάγει ήδη έρευνα κατά της gazprom για αντιμονοπωλιακή πολιτική. αυτή η έκθεση μπορεί να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήματα. από την άλλη πλευρά όμως κύριε επίτροπε μην ξεχνάμε ότι η ενέργεια και οι ενεργειακές σχέσεις απαιτούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα. ελπίζουμε ότι ο νέος μηχανισμός δεν θα διαταράξει υπάρχουσες καλές ενεργειακές καταστάσεις και σχέσεις των κρατών μελών με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσαβέλα. Και τώρα έχουμε τους λοιπούς ομιλητές με τον κύριο Φράνκο πρώτο για να Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Κάρινς, για την πολύ δύσκολη αυτή έκθεση μέσα στα πλαίσια του ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Έτσι θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή την απόφαση της Επιτροπής και χαιρόμαστε γι' αυτό. Προχωρεί η Ευρώπη, η κοινή Ευρώπη της ενέργειας και από διαφορετικής ε, πλευράς βρισκόμαστε σε κατάσταση εξάρτησης έναντι ορισμένων χωρών προμηθευτριών. Γι' αυτό θα πρέπει να εκπονήσουμε μια δική μας στρατηγική και μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει πληροφορίες σε σχέση με τις συμφωνίες ενεργειακού χαρακτήρα, ιδιαίτερα όσον αφορά την επικουρικότητα. Αυτό αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας και να μπορούμε να προτρέχουμε ως προς τις ανάγκες μας εφοδιασμού. Χαίρομαι γιατί δεν δημιουργούνται δεσμεύσεις μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων σε μια εποχή κρίσης και ανταγωνισμού και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει προστασία των ε, ιδιωτικών συμβάσεων. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ. Κύριε Φράνκο, κύριο Μπαλτσίτης, παρακαλώ για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ δυστυχώς. Κύριος Τζουρ, και ένα μισή λεπτό. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos az Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η προμήθεια ενέργεια των περισσότερων των ε, μελών ε, εξασφαλίζεται μέσω συμβάσεων διεθνών με τρίτα κράτη. Αυτές οι συμβάσεις όμω. δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονό ότι είμαστε η μεγαλύτερη αγορά ε, ενέργειας φυσικού βρισκόμαστε σε έναν άνισο αγώνα. Ε, τα ελαφρά βαρύ είμαστε εμείς, έναντι των βαρέων βαρών των ε, ενεργειακών μας εταίρων. Και έτσι, προφανώς, τα βαρέα βάρη βγάζουν νοκάουτ τα ελαφρά βάρη. Έτσι λοιπόν, η κοινοποίηση πληροφοριών, ε, η δημοσιοποίηση του σε κοινοτικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο θα μας ενισχύσει, θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε το ειδικό μας βάρος και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε οι καλύτερες συνθήκες για τις ε, συμφωνίες που θα συνάπτουμε ε, στον τομέα της ενέργειας. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν το ζητούν οι κυβερνήσεις να συμμετέχει και ενεργά στις διαπραγματεύσεις αυτές. Και ευχαριστώ, συγχαίρω δε και τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσικάου παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη-μέλη ώστε να έχουν πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές έτσι ώστε να έχουμε απρόσκοπτη μεταφορά ενέργειας. Μιλάμε για, τον, για την ενεργειακή ασφάλεια, για την ασφάλεια εφοδιασμού που μας απασχολεί πολύ σοβαρά και μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Επειδή θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα η ενεργειακή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να δούμε πώς θα, πώς θα οριστούν οι διακυβερνητικές συμφωνίες. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές από την Κομισιόν έτσι ώστε να τηρείται το νομοθετικό πλαίσιο η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και, και η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Γι' αυτό αυτό θα πρέπει να δώσουμε, να υπάρξει τεχνική αρρωγή από την Επιτροπή μέσα στα πλαίσια της ε, διακυβερνητικής ε, συνεργασίας. Ευχαριστώ την κυρία Τσικάου. Η κυρία Γιόρντον για 1,5 λεπτό. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εσωτερικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού ε, αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και ε, φυσικού αερίου έχει μεγάλη σημασία γιατί δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει συμφωνία για το πώς θα ε, λειτουργήσουμε. Μιλάμε για μια προστιθέμενη αξία η οποία, την οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δημιουργώντας και ορίζοντας αυτή την πολιτική. Επίσης έχει μεγάλη σημασία το πώς ε, οι αρχές αυτές θα μεταφερθούν και θα ενσωματωθούν σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Μιλάμε για μεταφορά εθνικής ευθύνης και αρμοδιοτήτων, κάτι το οποίο δεν επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Αυτό αφορά και το έγγραφο το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Αν και μιλάμε για τη σύσταση ενός μηχανισμού και όχι για τον έλεγχο καθεαυτό των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, το νομοθετικό κείμενο είναι αρκετά αποδυναμωμένο αλλά εν πάση περιπτώσει θα οδηγήσει στην εποπτεία της αγοράς ενέργειας. Στο μέλλον αυτός ο μηχανισμός θα αναβαθμιστεί εάν χρειαστεί. Γι' αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και επίγον να εγκρίνουμε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα μισή λεπτό, κύριο Κομισάριο. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κάρινς για τις διαπραγματεύσεις, τις επίπονες διαπραγματεύσεις με αποτέλεσμα αυτό το θετικό έγγραφο και νομίζω ότι έτσι θα δημιουργηθεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο για την εξωτερική μας πολιτική ενέργειας. Έτσι προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και στον τομέα της ενέργειας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την κοινή προσπάθεια και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες και γιατί ενέκρινε τις ε, διακυβερνητικές συμφωνίες και τις ενέταξε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη Συμφωνία Ανταλλαγής Πληροφοριών, πώς θα εξελιχθεί και ελπίζω να εξελιχθεί θετικά. Και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια των διακυβερνητικών συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας και θα ληφθεί υπόψη και η εξωτερική διάσταση της αγοράς ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Καρβάλιο. Ο κύριος Μπένσεν για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να συνεννοηθούν σωστά με την Gazprom στην Ρωσία. Ξέρουμε ότι η Gazprom έχει πολύ στενό σύνδεσμο με την πολιτική εξουσία της Ρωσίας, οπότε η επικοινωνία μαζί της είναι δύσκολη. Οι πρακτικές της Gazprom υπονομεύουν την εσωτερική αγορά και δεν επιτρέπουν να υπάρχει η διαφάνεια η οποία απαιτείται. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει ανάξι. Θα πρέπει το εμπόριο του φυσικού αερίου να λειτουργήσει σύμφωνα με τους σωστούς κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Ζητώ παρόλα αυτά τα μέλη να υπερψηφίσουν τη συμφωνία γιατί έχουμε και μια δυνατότητα ενδιάμεσης αναθεώρησης σε τρία χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Μπέντσελ. Ενάμιση λεπτό Μαρτσίνκεβιτς. Ευχαριστώ Επίτροπε. Η κρίση που είχαμε ζήσει με το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια έδειξε το πόσο τρωτή είναι η Ευρώπη. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για να ενισχυθεί η ασφάλεια της προμήθειας φυσικού αερίου δεν έχουν επαρκέσει. Έχουν πάντως υπάρξει κάποια μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο περισσότερο τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς απαιτείται καλύτερη ενημέρωση, απαιτείται καλύτερη πληροφόρηση. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Πολωνία και τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη και έκανε ορισμένες παρατηρήσεις για κάποιους όρους, τους οποίους είχαν επιβάλει οι προμηθευτές μας. Η Πολωνία είναι μια από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει στην διάθεσή της θα έλεγα ένα αρκετά αποδοτικό ανταλλακτικό μηχανισμό. Έχουμε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διεθνείς συμφωνίες τις οποίες συνάπτουμε σαν χώρα. Και τώρα διαπραγματευόμεθα επίσης κάποιες προμήθειες από την περιοχή της Κασπίας τις οποίες επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αγορά, η πολωνική λοιπόν δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από ανεύθυνες αποφάσεις. Γι' αυτό πρέπει να είναι σωστή η ενημέρωση και η επικοινωνία και να είναι ενήμερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Μαρτσίνκεβιτς. 1,5 λεπτό μέτσαρος. Κύριε Επιτροπέ, Κύριε Πρόεδρε, για την ανάπτυξη τη ε, βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ασφαλέ ενεργειακό περιβάλλον, σταθερέ προμήθειε ενέργεια. Αξιόπιστη λοιπόν προμήθεια ενέργεια μπορούμε να εξασφαλίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο εάν έχουμε μια ενιαία αγορά ενέργεια. Στην πρόταση αυτή μέτρων ε, πολλά κράτη που παρέχουν ή μεταφέρουν ενέργεια ε, μπορούν να ξεφύγουν από τους ελέγχους και μπορούν να ξεφύγουν από τους ελέγχους, μπορούν να ε, έχουν να υποστούν καλύτερους ελέγχους. Με την κρίση στο φυσικό αέριο το 2009 ε, ελέγχθηκε η αξιοπιστία των συστημάτων μας για την προμήθεια ενέργειας. Και έτσι για να έχουμε καλύτερες ε, τιμές για τον Ευρωπαίο καταναλωτή πρέπει να προβούμε σε συμφωνίες οι οποίες θα λειτουργούν κατά τρόπον σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο συμφωνίες με τρίτα κράτη οι οποίες θα λειτουργούν με βάση τους όρους της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι ο στόχος μιας ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να καλύψει ελλείψεις και διακυμάνσεις στην προμήθεια ενέργειας. Από την εμπειρία που έχουμε διαπιστώνουμε ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν τα κράτη-μέλη με τρίτες χώρες μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις σημαντικά και να βελτιώσει τις συνθήκες των συμφωνιών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μέσσερος και τώρα έχουμε τη δικασία Καρστιάη. Η κυρία Μπασέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη εξαρτάται από, εισαγωγές, από την εισαγωγή ενέργειας και μιλάμε για ένα ποσό 400 δις ευρώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό τον ευάλωτο τομέα, γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό μας. Θα πρέπει λοιπόν ο, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού να μας απασχολήσει μέσα στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής. Εμείς ε, βρισκόμαστε σε προνομιακή θέση και από γεωγραφικής και από γεωπολιτικής ε, πλευράς, διότι η Μαύρη Θάλασσα μπορεί να εξασφαλίσει τον ανεφοδιασμό μέσα στα πλαίσια ε, πολιτικών, περιφερειακών και οικονομικών μπλοκ. Ε, η χώρα μου υποστηρίζει σχέδια όπως ε, τον αγωγό Ναμποκο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον ε, εφοδιασμό μας από τις γείτονες χώρες. Ευχαριστώ πολύ και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καρίνη, συγχαρητήρια για την έκθεσή σας. Ήταν πολύ ορθολογική. Κύριε Επίτροπε, έχω μία ερώτηση σε αυτή τη διαδικασία ε, της εξέτασης των διακρατικών συμφωνιών η υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων της Επιτροπής θα παίζει καθοριστικό ρόλο γιατί θεωρώ ότι η ενέργεια θα πρέπει να είναι εκτός κανόνων εξωτερικής πολιτικής. Η ενέργεια έχει διάρκεια μεγάλη και προβλεψιμότητα την οποία οι εξωτερικές σχέσεις δεν έχουν. Ευχαριστώ. Κύριε Τζαβέλα, σας ευχαριστώ θερμά και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση, αλλά θα απαντήσει βέβαια, μάλλον για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Πίτροπο για να απαντήσει την κυρία Τζαβέλα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Βουλευτή. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη από όλε τι ομάδε εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κοινό ο στόχο να ενώσουμε τι δυνάμει μα και να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Στην αγορά αλλά και την προμήθεια ε, πηγών ενέργειας, πρωτογενών πηγών ενέργειας, θέλουμε περισσότερη διαφάνεια, ανταγωνισμό και βελτίωση των συμφωνιών που συνάπτονται με, τις, ε, με την υποστήριξη και τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και για τις επικρίσεις για την λίγο επικοδομητική στάση του Συμβουλίου γιατί υπήρξαν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής με μια κοινή συνεργασία, οι οποίες όμως απερίφθησαν από πλευράς του Συμβουλίου στην ουσία, έστω και αν στα λόγια το δεχόταν, απέριπτε τις προτάσεις συγκεκριμένε Ευρωπαϊκής επιτροπή. Πάντω ήταν σωστό ότι καταλήγουμε στο συμπέρασμα στο οποίο έχουμε έρθει σήμερα, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε τίποτα. Θα έπρεπε δηλαδή να ξεκινήσουμε από το μήτε δεν τις συζητήσεις. Έχουμε ήδη προχωρήσει κάποια μικρά βήματα στην υπόθεση αυτή. Έχουμε βάλει μερικά τούβλα στο δρόμο αυτόν και έχουμε κάπως προχωρήσει τις σχέσεις Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή από κοινού έχουμε βρει κάποιες λύσεις. Θα τις υλοποιήσουμε, στην πράξη θα ελέγξουμε, θα επαληθεύσουμε την υλοποίησή τους και στα δύο-τρία χρόνια που θα έρθουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαληθεύσει το πώς λειτουργεί αυτή η εξωτερική στρατηγική για την ενέργεια για να χαράξει το επόμενο και βαθύτερο βήμα στο δρόμο αυτόν. Εσείς ε, κυρία Τζαβέλα αναφερθήκατε στην ερώτησή σας στο κατά πόσον, στο πώς μάλλον η ενεργειακή πολιτική αλλά ειδικότερα, αλλά και η εξωτερική πολιτική γενικότερα μπορούν να αναπτυχθούν στον τομέα αυτών. Καταρχάς, η συνάδελφος Λέντι Άστον και εγώ έχουμε εξαιρετική σχέση και συνεργασία, την αναπτύσσουμε συνεχώς. Και όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, η ενεργειακή πολιτική έχει προτεραιότητα, όταν πρόκειται δηλαδή για τις σχέσεις μας με τρίτα κράτη, χωρίς εξαιρέσεις. Πάντοτε, δηλαδή, για λόγους ενεργειακής πολιτικής ε, δεν προτιμούμε να επιβάλλουμε μποϊκοτάζ στις εισαγωγές του πετρελαίου από το Ιράν για λόγους ενεργειακής πολιτικής. Και είναι μεγάλο ε, εξαγωγέα στο Ιράν. Μέχρι 30% είναι η εξάρτηση τη Ελλάδα αλλά και τη Ισπανία για τι εισαγωγέ του σε πετρέλαιο από το Ιράν. Όταν όμω έχουμε να κάνουμε μια ενιαία, μια αποφασιστική πολιτική και μια συνεπή πολιτική, τότε για λόγους όχι ενεργειακής πολιτικής αλλά για λόγους γενικής πολιτικής πρέπει να προχωρήσουμε και στο μποϊκοτάζ. Τότε θα πρέπει να το δεχθούμε. Και τότε η πολιτική ασφάλειας, η πολιτική ενέργειας και η πολιτική εξωτερική, η γενική πολιτική εξωτερικών σχέσεων συνεργάζονται και δίνουν λύσεις. Έχουμε συμφέροντα στην ενεργειακή πολιτική, την ειδική εξωτερική ενεργειακή πολιτική που δεν ε, μπορούν να υπαχθούν στη γενική εξωτερική πολιτική. Για το θέμα του Ναμπούκο που αναφέρατε επίσης και για το πώς αντιμετωπίζουμε την αναζήτηση νέων πηγών. Το 2018 πιστεύω μπορούμε να αναμένουμε αξιόλογες ποσότητες πετρελαίου από το Αζερβαϊτζάν και έτσι θα έχουμε μια νέα πηγή πέραν της Ρωσίας, πέραν της Νορβηγίας, πέραν της Αλγερίας και άλλων ε, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κάτω χώρες πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Με την ε, προοπτική για το Ναμπούκο, το Δυτικό Ναμπούκο, το Τάναπ και άλλα μέσα στου επόμενου εννέα μήνε περίπου, πιστεύω ότι θα μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Τώρα, εάν θα έχουμε μόνο από το Αζερβαϊτζάν φυσικό αέριο, αλλά ενδεχομένω και από το Τουρκμενιστάν ή και το Ιράκ, με τον ε, νότιο διάδρομο, τον South Corridor, εάν αυτό μετατραπεί δηλαδή σε ένα πραγματικό διάδρομο για το φυσικό αέριο, αντίστοιχο με αυτών των σχέσεων που έχουμε εδώ και δεκαετίες με την Ορβηγία, τη Ρωσία και την Αλγερία. Θα το δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Έτσιγκερ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο κύριος Κάνης έχει το λόγο, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, ιδιαίτερα του Σκιώδης. Καταφέραμε ό,τι το καλύτερο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δανέζικη Προεδρία καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνοψίζοντας, θα πρέπει να θυμόμαστε το βασικό μας μέλημα ως πολιτικών σε αυτό το τομέα. Μας ενδιαφέρει ο καταναλωτής και η τιμή της ενέργειας. Οι τιμές θα πρέπει να είναι χαμηλότερες και πιο δίκες. Το έγγραφο αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα που δημιουργεί μηχανισμούς ανταλλαγής απόψεων και ορίζει μια νομοθετική βάση για την μελλοντική κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Πολλοί επικρίνουν, πολλοί μας επικρίνουν που θέλουν περισσότερα, θέλουν ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο, μάλλον ένα τέλειο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βελτίωση των νόμων μπορεί να επιτευχθεί βεβαίως, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η σωστή βάση, δηλαδή να υπάρχει μια σωστή ρύθμιση. Ας θεωρήσουμε αυτό ως ένα σημείο εκκίνησης, ως ένα πετραδάκι για το μελλοντικό μας οικοδόμημα. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες και θα ήθελα να σας καλέσω να ψηφίσετε υπέρ της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ κύριε Καρίντς. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 και τώρα έχουμε από την ομάδα των συγχωριστών και Δημοκρατών ένα αίτημα για, ορισμό, για διορισμό μελών σε επιτροπές που κατατίθενται στα πρακτικά ανακοινώνονται μέχρι τις εκκρίσεις των